Seance on Direct. Δεύτερη ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές της Λιθουανίας κοινοποίησαν στο Κοινοβούλιο την ε, εκλογή της συναδέλφου Τζουστίνα Βιτκαουσκάιτε ω ε, ως αντικαταστάτρια του κυρίου Βίκτορ Ουσπάσκης ε, με ισχύ από 21 Νοεμβρίου 2012. Οι αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας ανακοίνωσαν στο Κοινοβούλιο την επιλογή της κυρίας Μόνικα Χάνς Πανιωτόβα ως αντικαταστάτριας του κυρίου Στέφανοφ Στογιάνοφ με ισχύ από 6 Δεκεμβρίου του 2012. Καλωσορίζω τους καινούριου συναδέλφους μας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού ε, έως ότου επαληθευθεί η εντολή τους ε, και δεν υπάρχει αμφισβήτηση η Τζουστίνα Βίκτκα Σκάιτε και η Μόνικα Χάνης Παναγιωτόβα ε, έχουν πλήρη δικαιώματα στο Κοινοβούλιο και στα όργανα του ε, εφόσον έχουν δηλώσει ότι δεν ε, έχουν καθήκοντα ε, μη συμβατά με αυτά του Ευρωβουλευτή. Τρίτη ανακοίνωση. Οι αρμόδιε γαλλικέ αρχέ διαβίβασαν στο Κοινοβούλιο το αίτημα άρση τη κοινοβουλευτική ασυλία τη κυρία Μαρή Λεπέν. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφο 2 του κανονισμού, το αίτημα αυτό παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή, δηλαδή στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.